τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης και τα έγγραφα που έχουν εγκριθεί είναι ήδη διαθέσιμα. Πρώτο θέμα της ε, ημερήσιας διάταξης είναι